Θα ήθελα τώρα να περάσω στην ημερήσια διάταξη. Τα πρακτικά της ε, συνεδρίασης της 17ης ε, Δεκεμβρίου είναι στην διάθεσή σας. Έχετε κάποια παρατήρηση? Αν όχι, εγκρίνονται. Να σας